Buon Σας καλησπερίζω για μια ακόμη φορά όλους. να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας, τον Τζέρι Μπράουν, κυβερνήτη της πολιτείας της Καλιφόρνια. Πήρε χθε στην μέρος στην διάσκεψη υψηλού επίπεδου για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας και σήμερα τον προσκαλέσαμε να πάρει μέρος στην συνάντηση, στην διάσκεψη των Προέδρων Πολιτικών Ομάδων διευρυμένη και με άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που το επιθυμούν. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μας να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με έναν Αμερικανό ηγέτη, μια χώρα την οποία θεωρούμε τον βασικό μας διεθνή συνομιλητή, τον κυβερνήτη μιας πάρα πολύ σημαντικής πολιτείας των ΗΠΑ, έναν πρωταγωνιστή της Αμερικανικής πολιτικής, η συζήτηση θα γίνει ως εξή μετά από μια παρουσίαση την οποία θα κάνει ο κυβερνήτης για 8 λεπτά θα πάρουν τον λόγο οι εκπρόσωποι των διαφόρων πολιτικών ομάδων θα θέσουν ίσως ερωτήσεις και ο κύριος Μπράουν θα κλείσει τη συζήτηση με μια παρέμβαση σύντομη. Είμαστε σχετικά ευέλικτοι ε, στον χρόνο, αλλά αγαπητέ κυβερνήτα, δυστυχώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τα άλλα τα κοινοβούλια. Eh, Οκτώ λεπτά πράγματι είναι λίγα για τη σημασία που θα έχουν οι συζητήσεις μας, αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να προσπαθήσετε και αν τα καταφέρετε. Λοιπόν, έχετε το λόγο αφού σας παρουσίασα πλέον. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στη συζήτηση. Νομίζω πως θα είναι επικοδομητική. Γιατί είμαι εδώ στην Ευρώπη σήμερα. Για να παρακολουθήσω, να συμμετάσχω στην COP23 για να προωθήσουμε τους στόχους της εφιούς ε, και δραστικής δράσης για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Καλιφόρνια είναι πιο ισχυρή από, πολλά, αλλά, από πολλές άλλες πολιτείες. Αλλά η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια απειλή. Χρειάζεται και παγκόσμια δράση. Αλλά αυτή η δράση βεβαίως πρέπει να αναλυφθεί από άτομα, από πολιτείες, από περιφέρειες, από κράτη. Χρειάζεται πραγματική κινητοποίηση των κρατών του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολλά οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει, έχουν αποχωρήσει, αλλά πιστεύω ότι θα επανέλθουν τα επόμενα χρόνια. Αλλά διάφορες πολιτείες και άλλες δικαιοδοσίες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια τους. Έχουμε τώρα μια ευρεία συμμαχία όπου συμμετέχουν περίπου 190 πολιτείες και επαρχίες που εκπροσωπούν το 1 τρίτο του παραγωγικού δυναμικού σε όρους ΑΕΠ του πλανήτη πάνω από ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. Είναι μια ισχυρή λοιπόν συμμαχία, μια ισχυρή δέσμευση για να αντιμετωπιστεί αυτή η υπαρξιακή απειλή. Πολλές απειλές είναι στην ουσία. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο ευάλωτες ε, οι χρηματοπιστωτικές δομές από όσο θα θέλαμε. Το πυρηνικό θέμα γίνεται όλο και πιο απειλητικό. Αλλά παρόλα αυτά η κλιματική αλλαγή είναι επίσης από τις ε, κύριες απειλές και γι' αυτό είμαι μεταξύ σας εδώ στην Ευρώπη σήμερα. Ξέρω, γιατί είδα πώς εξελίχθηκε το θέμα στην Καλιφόρνια, ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Έχουμε αναλάβει δράση για να μειώσουμε τις εκπομπές ε, άνθρακα θέλουμε να κατέβουμε στο επίπεδο του 1990, αλλά και τότε ήμασταν υψηλά. Η Καλιφόρνια ήταν περίπου στους 12 τόνους ανακάτοικο αερίων θερμοκηπίου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε συνολικά είναι στους 18-19 τόνους, άρα πολλά μένουν να κάνουμε. Αλλά έχουμε κάνει ορισμένα πράγματα στις προδιαγραφές για τις εκπομπές των αυτοκινήτων. Έχουμε αυτή τη στιγμή 300.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και θέλουμε να φτάσουμε στο 1,5 εκατομμύριο στα επόμενα 7 χρόνια έχουμε προδιαγραφές για τις ανανεώσιμες είμαστε περίπου στο 30% και θεωρούμε ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε φτάσει στο 50%. Επίσης έχουμε και τη λεγόμενη προδιαγραφή ότι η βενζίνη που χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει 10% λιγότερες, να παράγει 10% λιγότερες εκπομπές από την ε, ε, μέση εκπομπή καυσαρίων της βενζίνης. Είναι πολύ τεχνική αυτή η προδιαγραφή και απαιτείται από τις εταιρείε είτε να χρησιμοποιούν δύο καύσιμα ή την, ε, να χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες ή να πληρώνουν για το δικαίωμα να μην το κάνουν. Και επίσης έχουμε πολύ σημαντικές προδιαγραφές για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για τα κτίρια και για τις ηλεκτρικές συσκευές και έχουμε αναθεω... αναθεωρήσει γενικά τις προδιαγραφές μας, τις προδιαγραφές μας μέχρι το 2030. Με πολύ ευρία πλειοψηφία, δύο τρίτα ε, στη... στο τοπικό μας κοινοβούλιο και 8 ρεπουμπλικανοί από τους 120 ψήφισαν και αυτοί μαζί μας. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ποτέ πουθενά αλλού στην Αμερική δεν έχουν υπάρξει τόσο, ρεπουμπλικανοί, τόσο πολλοί ρεπουμπλικανοί που να ψηφίζουν για κλιματική δράση. Υποθέτω ότι αυτός όμως ήταν και ο λόγος που ο ρεπουμπλικανός ηγέτης που προκάλεσε αυτήν την ψήφο των συναδέλφων του υπέρ της κλιματικής αλλαγής τελικά ε, απορρίφθηκε και αποσύρθηκε απορρίφθηκε από τις τοπικές οργανώσεις ε, ρεπουμπλικανών. Ξέρετε, στη χώρα μου υπάρχει βαθιά ε, δυσπιστία και απόρριψη της επιστημονικής σκέψης που λέει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λειτουργεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, άρα αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις στην Καλιφόρνια, όπως και στην υπόλοιπη χώρα. 13-14 άλλες πολιτείες συνεργάζονται μαζί μας σε διάφορα επίπεδα ε, για κλιματική δράση. Και νομίζω ότι θα προσθεθούν και άλλες. Αλλά είναι τόσο επικίνδυνη αυτή η απειλή και τόσο τεράστια η αντίδραση που χρειάζεται που η μόνη πιθανότητα να επιτύχουμε είναι να αυξηθεί κατά πολύ η συνειδητοποίηση, να δεσμευτούν πολύ περισσότεροι και ε, να δεσμευτεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα κράτη και περιοχές. Η Κίνα επίσης, που μέχρι στιγμής ε, είναι ιδιαίτερα αρνητική, η Ινδία, η Αφρική, γιατί όλοι θα επηρεαστούν. Άρα όλοι πρέπει να αντιδράσουν. Αλλά μόνο όσοι είναι ε, θέση που να τους επιτρέπει να αντιδράσουν μπορούν να αναλάβουν αποφασιστική δράση. Οπότε σας καλώ να αναλάβετε περαιτέρω δράση ενώ εγώ προσπαθώ στην δική μου χώρα να αυξήσω την συνειδητοποίηση. Δεν έχουμε ακόμη αντιμετωπίσει επαρκώς τον κίνδυνο. Και μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο καμπής στην αύξηση της θερμοκρασίας και αν το υπερβούμε τότε θα υπάρξουν ε, αποτελέσματα που δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στο κλίμα και σε μεταναστευτικές ροές. Και ίσως σε ορισμένες περιοχές αυτό να συμβεί σύντομα. Δεν μπορούμε λοιπόν να εφησυχάζουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πολύ εφησυχασμό στην περιοχή μου τουλάχιστον, στην χώρα μου. Θα πάω λοιπόν στο COP23, ούτως ώστε μαζί με άλλα κράτη, άλλες πολιτείες, άλλες περιφέρειες το, όπως το Κεμπέκ και το Ράριο, τα, οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Ουάσιγκτον, του Όρεγκον και περιοχές της Κίνας, της Ευρώπης, της ε, Νότιας Αμερικής. Περιοχές παντού στον κόσμο προσπαθούν να συνεργαστούν από τη βάση προς τα πάνω, ούτω ώστε να προωθήσουμε την κλιματική αλλαγή για να έχουμε αποτελεσματική δράση. Γι' αυτό είμαι εδώ για να συζητήσω, να ακούσω τις ιδέες σας, αλλά οι δικές μου ιδέες είναι απλές. Ο κίνδυνος είναι θεμελιώδης. Θα αλλάξει ο πολιτισμός μας. Και δεν απέχει δεκαετίες. Είναι πολύ κοντύτερα από ό,τι νομίζετε. Και δεν θα επιτύχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνδυνο εάν δεν δράσουμε τάχιστα και σε βάθος. Με βιώσιμο τρόπο πρέπει να πείσουμε τους συμπολίτες μας και πρέπει να δράσουμε παγκόσμια. Αυτά ήθελα να σας πω και με χαρά να ακούσω τις ερωτήσεις σας και να συζητήσουμε το θέμα αυτό όποιο τρόπο θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπράουν, κυβερνήτα Μπράουν που σεβαστήκατε απόλυτα και το χρόνο σας. Χαίρομαι ως Προεδρεύων. Τώρα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η Μάιριτ Μαγκίνες, πρώτη αντιπρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ελπίζω να ικανοποιηθείτε και από τη δική μου επίδοση σχετικά με το χρόνο. Ευχαριστώ κυβερνήτα για μια πραγματικά ξεκάθαρη παρουσίαση. Ήταν ενδιαφέρουσε οι παρατηρήσει σας ότι στην ουσία είπατε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σε σχέση με το Παρίσι έχουν αποστασιοποιηθεί και δεν μετέχουν. Και είπατε επίσης και τη σημασία έχει αυτό που κάνει ο κάθε πολίτης και τα μεμονωμένα και οι μεμονωμένες οντότητες όπως οι πολιτείες. Είναι σαφές ότι και εκεί μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ενδιαφέροντα τα σχόλια που κάνατε και στην πόλη του Βατικανού. Θα μπορούσατε να επανέλθετε λίγο σε αυτά, να πω στους συναδέλφους ότι μιλήσατε σε ένα συμπόσιο για το περιβάλλον στο Βατικανό και είπατε ότι το θέμα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του περιβάλλοντος απαιτεί όχι μόνο επιστημονικές προσπάθειες αλλά ακόμα και προσπάθειες σε επίπεδο πίστης, θρησκείας. Ε, πράγματι εμείς ε, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με το περιβάλλον είναι να μην είμαστε αδρανείς, να μην είμαστε αδιάφοροι, να μην είμαστε απαθείς και αντίθετα να είμαστε ενθουσιώδεις και επίμονοι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα πείσουμε από εδώ και πέρα αυτούς οι οποίοι κατανοούν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το κλίμα και να οδηγήσουμε σε αλλαγές οι οποίες θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν, ζουν και εργάζονται. Ε, μπορούμε εμείς ε, να πείσουμε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο έτσι ώστε ο κόσμος να στραφεί προς μια κατεύθυνση την οποία εμείς θεωρούμε ευταία και ε, θα πρέπει να την ακολουθήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αναλάβει σοβαρότατες υποχρεώσεις, αλλά απαιτείται από μεμονωμένους τομείς όπως ο αγροτικός τομέας να μην ανησυχεί όσο ανησυχεί σήμερα. Θεωρεί η Γεωργία ότι τη ζητείται να γίνει περισσότερα, να κάνει περισσότερα από ό,τι άλλοι τομεί και ιδιαίτερα στον τομέα τη κτηνοτροφίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβουμε δράσει που θα έχουν σημαντικέ επιπτώσει. Το ίδιο και στι οικοδομέ, το ίδιο και στι μεταφορέ. Πάντως όταν κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός υπάρχουν δυστυχώς δυνάμεις που μας οδηγούν πίσω έστω και κατά μισό βήμα. Η σοφία λοιπόν και η γνώση σας μας είναι απαραίτητες έτσι ώστε να εμείνουμε στον δρόμο που ακολουθούμε. Όταν αναφερθήκατε στο Βατικανό λοιπόν για αυτήν την ανθρώπινη αδράνεια, την υπερβολική φιλοδοξία ε, και τον αρνητικό τρόπο που βλέπει τις κλιματολογικές αλλαγές. Πώς θα αλλάξουμε αυτά τα αισθήματα, ιδιαίτερα στον αναπτυγμένο κόσμο. Τους πολίτες που δεν είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν λίγο τη βολή τους για το κοινό καλό. Νομίζω ότι αν μας απαντήσετε σε αυτό θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κλίματος με τον σωστό τρόπο που εσείς γνωρίζετε. Επιστρέφοντας τώρα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στις Ηνωμένε Πολιτείε, ένα από τα σχόλια τα οποία ακούμε από τους Αμερικανούς είναι ότι εμεί θα πρέπει να δράσουμε ενώ άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να σχολιάσετε. Και σε σχέση τώρα με την προσπάθεια να δώσουμε μάχες από τα κάτω προς τα πάνω, από τη βάση προς τα πάνω. Πολύ ενδιαφέρον πώς αναπτύσσεται μια τέτοια κίνηση στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ένα τελευταίο σημείο που θέσατε είναι εύκολο να κάνει κανείς κάτι το μικρό αν είστε από τους πιο σημαντικούς σε εισαγωγικά εκπομπής. Λοιπόν, πώς μπορούμε να πείσουμε ε, τους φτωχότερους, τους μετανάστες, ε, τους ασθενέστερους ότι τα συμφέροντά τους δεν θα αγνοηθούν στα πλαίσια αυτή της συζήτηση. Η κυρία Βαν Μπρέμπτεξ, των Σοσιαλιστών και Δημοκράτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον κυβερνήτη Μπράουν στη συνεδρίασή μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις στην παρούσα συνεδρίαση. Επιτρέψτε μου να αρχίσω παραθέτω τον Μπέντζαμιν Μπάρμπερ που είναι γνωστός λοιπόν βέβαια πανεπιστημιακός τον οποίο γνώρισα καλά και ήταν καλός μου φίλος και έγραψε πολλά βιβλία και το πιο γνωστό του είχε τον τίτλο «Τι θα συνέβαινε αν οι δήμαρχοι κυβερνούσαν τον κόσμο». Γιατί ε, εσείς δεν είστε μόνο σήμερα ε, κυβερνήτη στην Καλιφόρνια, αλλά έχετε σπάσει και όλα τα ρεκόρ ε, ε, ε, ε ως κυβερνήτης, αλλά διατελέσατε και δήμαρχος της Όκλαντ. Άρα ο κόσμος θα ήταν καλύτερα, σε καλύτερη κατάσταση αν κυβερνούσαν οι δήμαρχοι γιατί εκείνοι είναι οι πολιτικοί που βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, γνωρίζουν τι σημαίνει στην πόλη τους και βλέπουν και ποιοι ε, πλήττονται σήμερα και ποιοι υποφέρουν. Παγκοσμίω, όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Παρατηρούμε ότι οι δήμαρχοι και άλλοι τοπικοί ε, άρχοντες αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή πόλεις, περιφέρειες, κράτη έχουν συμμαχήσει, όπως στη συμμαχία στην οποία αναφερθήκατε εσείς. Η Καλιφόρνα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Έχει αναλάβει μεγάλη δράση στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν είστε μόνο σημαντική πολιτεία αλλά και έκτη μεγαλύτερη οικονομία. Ε, εμείς συζητάμε αυτό τον καιρό για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλα καυσαέρια. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τεχνικές, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι... Ε, έχουμε υιοθετήσει κάτι ε, το οποίο κάνετε εσείς από το 1990 στο πρόγραμμα ZEF στην Καλιφόρνια με στόχο 1,5 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα ε, οχήματα μέχρι το 2025 και δώσει το καλό παράδειγμα και για την Ευρώπη. Ένα δεύτερο στοιχείο πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής είναι η κοινωνική διάσταση. Μήπω να το πω διαφορετικά, η κλιματική αλλαγή είναι κυρίως κοινωνικό ζήτημα σήμερα. Και είναι θέμα αναδιανομής. Αν δεν προσέξουμε. Αυτό θα εντείνει και τις ανισότητες και ε, τις συγκρούσεις και τις αβεβαιότητες και την ανασφάλεια. Για να συνεργαστούν όλοι θα πρέπει να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση και σωστή προς μια οικονομία επιλαγμένη από το διοξίδιο του άνθρακα. Καθόλου εύκολο δεν θα είναι αυτό. Όχι επειδή δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι και πώς θα φτάσουμε σε αυτούς, αλλά γιατί πολύ τυφλωνόμαστε από το φόβο μήπως χάσουμε προνόμια και εξουσία. Και ο μέσος ψηφοφόρος σήμερα ανησυχεί βαθύτατα για την αλλαγή στον πλανήτη αλλά και για την αλλαγή στην καθημερινή του ζωή. Και ποια είναι εδώ η δυσκολία. Ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης για να περάσουμε σε μια νέα οικονομία θα πρέπει να ε, συμμετέχουν όλοι και όχι μόνο κάποιοι εκλεκτοί και να γίνει μεν μετάβαση αλλά με προστασία για τον ε, κόσμο, για τους εργαζομένους για να έχουν αξιοπρεπή εργασία και αξιοπρεπή συνθήκες εργασίας. Και τέλος κυβερνήτα υπάρχει και κάποια ελπίδα γιατί όταν ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αποσυρθούν από ε, τη Συμφωνία των ε, Παρισίων κάποιοι φοβήθηκαν ότι θα μειωθεί η κάθε φιλοδοξία. Το αντίθετο συνέβη. Οι παγκόσμιοι ηγέτες και τα κοινοβούλια συσπηρώθηκαν στην προσπάθεια αυτή. Και θέλω πάλι να τονίσω το γεγονός ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές πόλεις και πολλές πολιτείες αντιδρούν. Ακόμα και αν κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον λέει το αντίθετο και λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα για μια κοινή αγορά για το διοξείδιο του άνθρακα δεν συζητάει με την Ευρώπη Ουάσιγκτον αλλά εσείς. Ερωτήσει τώρα για να κλείσω. Η πρώτη είναι γενικότερη. Αναφερθήκατε σε αυτό, κυβερνήτα. Πώ μπορούμε εμεί από την ευρωπαϊκή πρόπτικη να σα βοηθήσουμε για να σφυριλατήσετε τη Συμμαχία των προθύμων στι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αναλάβουν τις υποσχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, πολιτείες και οι πόλεις τώρα, αλλά τι γίνεται και με τις οικονομικές υποσχέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. The next speaker is Mrs. Stevens, in name of the Group. Εξ ονόματος της και Μεταρρυθμιστών, η κυρία Χέλγα Στέβενς. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπράουν, που βρήκατε χρόνο να συζητήσετε μαζί μας. Νομίζω ότι οι σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικές για να βρούμε λύσεις στα κοινά προβλήματα που μοιραζόμαστε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι το άλλο μου σπίτι. Εγώ ε, πήρα πτυχίο νομικής από τον Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια ε, και έζησα και ένα χρόνο στο Μισούρι, στο Σεντ Λούις. Η Καλιφόρνια είναι ένας χώρος γεμάτος δημιουργικότητα και φάνταστη δημιουργικότητα για το μέλλον. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν και η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστούν στα πιο σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε. Ποτέ οι προκλήσεις δεν ήταν τόσο μεγάλες αλλά και τόσο κοινέ. Απαιτείται φιλόδοξη συνεργασία διασυνοριακά, διασφαλίζοντας την εσωτερική και διεθνή ασφάλεια των πολιτών μας, αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή κρίση δημιουργώντας ισχυρούς και ελεύθερους εμπορικούς ε, δέσμους και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα και τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της αύξησης του διεθνούς πληθυσμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι ένα <clears throat> πρόβλημα το οποίο θα μπορούμε να αγνοούμε για πολύ καιρό για οικονομικούς λόγους θα πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε πράγματα για να προστατεύσουμε τις γενιές του μέλλοντος. Γι' αυτό σωστά υπογραμμίζεται τη σημασία του προβλήματος και γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως τη Συμφωνία των Παρισίων έτσι ώστε το μέλλον να μην εξαρτάται μόνο από τα συμφέροντα των επιχειρήσεων αλλά να στηρίζει μια οικονομία η οποία να μπορεί να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και στην αηφόρο ανάπτυξη να πείσουμε τους επενδυτές ότι αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Αν δεν τα καταφέρουμε η πολιτική μας θα αποτύχει. Η πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο μείγμα πραγματισμού και ουτοπικής σκέψης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα στον τομέα της βιομηχανίας υλικών για τις οικοδομές. Ε, υπάρχουν πολλά τα οποία έχετε κάνει, τα οποία είναι ενδιαφέροντα και για μας, όπως οι νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες έχετε προχωρήσει και είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει και τους γείτονές σας που το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με φιλόδοξο τρόπο αλλά να κάνουμε και τους απαραίτητους συμβιβασμούς. Πολλές φορές τα βήματα της προόδου είναι βήματα μικρά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι φιλοδοξίες μας είναι μικρές. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την ε, επιχειρηματικότητα και με τη βιομηχανία, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον βελτιώσιμο με αηφόρο τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ καλό το ότι είσαστε ανάμεσά μας σήμερα για να μοιραστείτε μαζί μας αυτά τα οποία κάνετε στην Καλιφόρνια, ιδιαίτερα σε σχέση με τα οικονομικά κίνητρα για πιο καθαρά αυτοκίνητα, ιδιωτικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία κτλ. Νομίζω ότι αυτά έχουν μια διάσταση όχι μόνο πολιτιακή ή εθνική, αλλά έχουν μια παγκόσμια διάσταση σε επίπεδο ΠΟΕ. Βέβαια η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Όπως είπατε στην επίσκεψή σας στο Πεκίνο, τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο και τίποτα δεν είναι και πιο σημαντικό. Να αποδείξουμε ότι οι χαμηλές εκπομπές είναι καλές για την επιχειρηματικότητα, καλές για το περιβάλλον, καλές για τους καταναλωτές οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι ευρωπαϊκές αξίες μοιράζονται αξίες, ιστορία και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλος. Η ασφάλεια και η οικονομία συμβιώνουν σε έναν παγκοσμιωμένο κόσμο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ λοιπόν και τίνατε χείρα φιλίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία μας στο μέλλον. η κυρία Μπίατζα για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κυβερνήτα που ήρθατε να μιλήσετε. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούσαμε ότι υπήρξε πολύ δημόσια ανάκτηση ε, λόγω του ότι αποχώρησαν οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, από την Συμφωνία των Παρισιών αλλά υπάρχει η ίδια ανάκτηση και καταγγελία ε, όταν γίνονται τόσες επιθέσεις κατά του περιβάλλοντος μας όταν καταστρέφονται τα δάση όταν κυνηγούν τα ζώα για τρόπεα όταν καταστρέφεται το περιβάλλον γύρω μας και βλέπουμε ότι σε διάφορα μέρη του κόσμου υπάρχει τεράστια απειλή κατά του περιβάλλοντος και το αμερικανικό και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας ε, του Περιβάλλοντος ε, έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιοχές ε, βοηθούν να αντιμετωπιστεί η λαθροθυρία κατά των ελεφάντων. Αλλά βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει περικόψει κατά πολύ τους πόρους για αυτά τα προγράμματα ακόμη και από το πρόγραμμα για την ε, προστασία των ελεφάντων της Αφρικής και της Ασίας. Και αυτές οι περικοπές γίνονται μια άθλια στιγμή, ιδιαίτερα για τους αφρικανικούς ελέφαντες γιατί θανατώνονται για το ε, ελεφαντόδοντο ε, με ρυθμό 1 κάθε 15 λεπτά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς η χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Ω κυβερνήτη τη Καλιφόρνια, πόσο προστατεύετε το τοπικό περιβάλλον μαζί με τις εκστρατείες σας για την κλιματική αλλαγή. Θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκή συνειδητοποίηση στο κοινό και στους νομοθέτες για την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος παντού. Όλοι αγαπάμε το φυσικό περιβάλλον, ε, την ε, άγρια φύση, αλλά πάντα περικόπτονται οι πόροι όταν πρόκειται για να προστατευτεί αυτό το τοπικό περιβάλλον. Γιατί νομίζετε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε κυβερνήτη. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ η κυρία Άνια Χάζεκαμπ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυβερνήτα Μπράουν. Είναι προνόμια να σας ακούμε. Να μιλάτε για τον τρόπο με τον οποίο εμπνέετε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή με πρωτοβουλίες για αλλαγή συμπεριφοράς. Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι απειλή ε, για ανθρώπους, ζώα, για κτίρια. Θέλουμε να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στους δύο βαθμούς Κελσίου. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι δεν κάνουμε αρκετά για να πετύχουμε το στόχο αυτό που έχουμε θέσει. Θα σας μιλήσω για τα αυτοκίνητα και δεν θα σας εκπλήξει το θέμα που είναι η βιομηχανική γεωργία. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία, από τη βιομηχανική γεωργία είναι μεγαλύτερες των μεταφορών είναι πολύ σημαντικό για την κλιματική αλλαγή και αν δεν δράσουμε τώρα θα χειροτερεύσει η κατάσταση. Πριν από 15 χρόνια είχαμε 15 δισεκατομμύρια ζώα σε εκτροφές, ενώ σήμερα έχουμε 24 δισεκατομμύρια εκτρεφόμενα ζώα. Δηλαδή έχουμε τριπλάσιο αριθμό ζώων εκτροφής ε, στον πλανήτη από ό,τι ανθρώπους. Και για να δώσουμε ζωοτροφές στα ζώα αυτά καλλιεργούμε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αν σταματήσουμε να παράγουμε ζωοτροφές και χρησιμοποιήσουμε ε, τα εδάφια αυτά για καλλιέργεια τροφίμων, ε, μπορούμε να έχουμε τροφή για 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Ενώ αν αρχίσουν οι Ινδοί να τρώνε κρέας κάθε μέρα και εμείς τέσσερις μέρες την εβδομάδα, ε, αυξάνουμε τις εκπομπές κατά 814 μεγατόνους. Άρα θα πρέπει να καταναλώνουμε λιγότερα ζωικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Κρέας. Παράδειγμα, αν καθένας στις Ηνωμένε Πολιτείες τρεις μέρες την εβδομάδα δεν ε, τρώει κρέας θα εξοικονομήσουμε εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου αντίστοιχες με όλη την παραγωγή ε, πετρελαίου ε, στον κόλπο του Μεξικού, 17% της συνολικής πετρελαιοπαραγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν στις Ηνωμένε Πολιτείες σταματήσουν οι πολίτες να καταναλώνουν κρέας έξι μέρες την εβδομάδα, θα εξοικονομήσουμε ε, εκπομπέ οξυδίου του άνθρακα και αερίων θερμοκηπίου ε, της πολιτείας της Καλιφόρνια, ε, της Σα σας έφερα δύο βιβλία σχετικά για να σας εμπνεύσουν στις διαπραγματεύσεις της COP23. Τι προτίθεστε να κάνετε λοιπόν για να επιταχύνετε τη μετάβαση σε μια διατροφή περισσότερο φυτική και λιγότερο ζωική. Ο κύριος Ζαντό, εξ ονόματος των Πρασίνων. Κύριε Κυβερνήτα, καλωσορίσατε ε, στις Βρυξέλλες, ε, καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρίσκεστε τώρα σε μια ιδιαίτερη κατάσταση εσείς που τελικά η οικονομία στην Καλιφόρνια είναι πιο σημαντική από πολλές εθνικές οικονομίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν συμμετέχετε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και αυτό με οδηγεί ε, στα εξή δύο σημεία για την COP23. Δύο κινδύνους θέλω να αναφέρω που θεωρώ σημαντικού αυτή τη στιγμή. Ισχύει η Συμφωνία των Παρισίων, αλλά αυτή τι σημαίνει. Τα εξή δύο. Ένα πολύ φιλόδοξο στόχο, 1,5 με 2 ε, βαθμού το πολύ στα τέλη ε, του αιώνα και τόσο το καλύτερο. Γιατί ασχολείται η επιστήμη με αυτά, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη μας είπαν ότι η Συμφωνία των Παρισίων σημαίνει και κάποιες ε, υποχρεώσεις από τα κράτη-μέλη που υπολείπονται πάρα πολύ. Άρα θα πρέπει να περάσουμε από την κλιματική διπλωματία με πάρα πολύ ωραία και μεγαλόστομα λόγια στην κλιματική δράση για να τηρούν τις υποσχέσεις τους και τις υποχρεώσεις τους οι χώρες, τα ενεχόμενα ε, μέλη στον Ερωτώ λοιπόν πώς θα εξασφαλίσουμε ακριβώς αυτή τη στάση. Στη δεκαετία του 90 ε, πολλές φορές τα κράτη ήταν πιο προχωρημένα από τις κοινωνίες. Τώρα σημαίνει το αντίθετο. Δεύτερη ερώτηση για την COP23. Η COP23 και οι διασκέψεις του ΟΗΕ κινδυνεύουν να γίνουν μία έκθεση ε, παρουσίασης ε, των επιχειρήσεων και των εταιριών που έχουν δράσει, των πολιτών που δρούν, των δήμων, των κοινοτήτων, των περιφερειών, των επαρχιών και τελικά ε, τα κράτη κρύβονται πίσω από τη δράση όλων αυτών των μη κυβερνητικών και μη κρατικών ε, φορέων για να αδρανήσουν. Και υπάρχει κίνδυνος, γιατί όταν τόσο πολύ επενούμε κάποιους δήμους, κάποιες εταιρείες και κάποιες επαρχίες και περιφέρειες, να χαλαρώσει η πίεση προς τα κράτη. Αλλά αν θέλουμε να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου θα πρέπει τα κράτη τα ίδια να δράσουν πολύ περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας. Έχετε την αίσθηση ότι καμιά φορά εσείς είστε ένα υποκατάστατο στη δράση των κρατών και για τα κράτη ένα άλοθη για την αδράνειά τους. Επόμενο ερώτημα. Για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ο πρόεδρος Ομπάμα ε, κατήργησε ε, ένα σχέδιο αγωγού ε, γιατί θεωρούσε ότι ήταν κλιματοκτόνος αυτό το μεγάλο έργο. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σταματήσει την εισαγωγή πετρελαίου, σχιστολιθικού αερίου και ε, ε, διαφόρων ε, πετρελαιούχων μάλλον ασφαλτούχων άμμων θεωρείτε σκόπιμο κάτι τέτοιο θα βοηθούσε Και τέλος, η Καλιφόρνια περισσότερο από την Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να αναπτύξει ένα οικονομικό μοντέλο που να βασίζεται ταυτόχρονα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και στην ψηφιακή οικονομία. Να έχει μια κλιματική οικονομία δηλαδή όπου τελικά οι νέες τεχνολογίες είναι σύμμαχοι της καθαρής ενέργειας ή της εξοικονόμησης ενέργειας με τη μείωση της κατανάλωσης. Θεωρείτε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να εξαχθεί στις υπόλοιπες Ηνωμένες Πολιτείες από την Καλιφόρνια και στην Ευρώπη στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας η κυρία Λούνγκρεν. Ο κύριος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φίντσο ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί και θα σας διαβάσω την ομιλία του. Κυβέρνητα Μπράουν, σας ευχαριστώ στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας, σας καλωσορίζω. Πριν από μερικές μέρες στη Ρώμη καλέσατε να γίνουν παγκόσμιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή λέγοντας ότι μικρή επίδραση έχει ο Τραμπ, αλλά νομίζω ότι πολλοί διαφωνούν. Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει πρώτα τα αμερικανικά συμφέροντα και πολλοί πιστεύουν ότι η αποχώρηση από τη Συμφωνία των Παρισίων ήταν σωστή πράξη. Πολλοί, όπως και εγώ, ε, υποστηρίζουμε το σκεπτικισμό για την κλιματική αλλαγή που προωθείται από τα πράσινα λόμπι. Εδώ στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει και άλλους στόχους για μείωση των εκπομπών. Ποτέ δεν τελειώνουν οι πολιτικές μας μας υποχρεώνουν να κάνουμε τρομερές επενδύσεις ε, που θα έχουν πολύ μικρά αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Για διάφορες δεκαετίες θα αυξάνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτές οι προσπάθειες που γίνονται στην ουσία μπορεί να στείλουν τις επιχειρήσεις που εκπέμπουν πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε περιοχές του κόσμου όπου θα είναι ακόμη υψηλότερη. Στην ουσία αντιμετωπίζουμε ένα υποθετικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σε πολλές δεκαετίες. Έχει άδικο, είναι άδικη η πολιτική αυτή και υπάρχει τρομερή υπερτίμηση. Η μικρή αλλαγή και αύξηση της θερμοκρασίας που έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο αιώνα είναι απόλυτα φυσιολογική και έχει να κάνει με τις κυκλικές αλλαγές που παρατηρούμε τα τελευταία 10.000 χρόνια. Είχαμε σε διάφορες ε, στιγμές ε, υψηλέ ε, και χαμηλέ θερμοκρασίε από την Ρωμαϊκή εποχή, το Μεσαίωνα κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο. Δεν χρειάζεται ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Βεβαίω, οι παγετώνε αυξάνονται στι περιόδου αύξηση θερμοκρασία, συγγνώμη, αύξηση μειώνονται τότε και αυξάνονται όταν κατεβαίνει θερμοκρασία. Και οι αριθμοί των πολικών αρκούδων ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Άνοδος ε, του επίπεδου της θάλασσας μα ανεβαίνει εδώ και 10.000 χρόνια. Και γενικά ε, η αύξηση του επίπεδου της θάλασσας μειώνεται τώρα. Και όλοι αυτοί που λένε ότι θα πληγούν διάφορα νησιά λένε ανοησίες. Οι περισσότεροι επιστήμονες, 97% συμφωνούν με αυτό. Έχει απόλυτα διαψευστεί αυτή η κινδυνολογία. Όλα αυτά λέγονται από μη επιστήμονε. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πολύ σημαντικές ε, συζητήσεις μεταξύ των ε, επιστημόνων για το αν υπάρχει όντως κλιματική αλλαγή. Ενώ η αρμόδια επιτροπή δεν είναι ανεξάρτητη. Είναι μια ομάδα που έχει λάβει εντολή να βρει στοιχεία που να ε, ενισχύσει να ενισχύουν την κλιματική ιστερία. Διάφορες βιομηχανίες από την ε, χαλιβουργία ε, μέχρι την φαρμακευτική βιομηχανία και τη χημική βιομηχανία υποφέρουν. Ε, ελπίζω κάποια στιγμή η χώρα μου να αποκτήσει τη δυνατότητα να έχει το πεπρωμένο στα χέρια της και να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό σχέδιο για την ενέργεια. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα τώρα, εσείς την έχετε μάλλον στις ΗΠΑ και θα, πρέπει να είστε είσαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ο κύριος Γουλφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κυβερνήτη Μπράουν. Είναι η πρώτη ευκαιρία που μου δίδεται να συζητήσω με ένα δημοκράτη κυβερνήτη. Είχα, με είχε ε, συναντηθεί με τον Μάικ Λί, τον Σκοτ Βόκερ και είχαν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένε Πολιτείες θα πρέπει να δράσουν στον τομέα του κλίματος. Πάντως είδατε η Ευρωπαϊκή Ένωση σας καλωσόρισε σήμερα γιατί συμφωνείτε μαζί της, είστε στην ε, και εσείς αφιερώσατε τη ζωή σας στην πολιτική αποκλειστικά, θέλετε να ξοδεύετε τα χρήματα των φορολογουμένων συνεχώς, θέλετε να υπάρχει συγκεντρωτικό κράτος και ταυτόχρονα διαφοροποιήστε από τις Ηνωμένε Πολιτείες και λέτε ότι οι ψηφοφόροι ψήφισαν την ε, Κυρία Κλίντον, συνεπώς έχετε μια πολιτεία διαφορετική από τις υπόλοιπες Ηνωμένε Πολιτείε με τέτοια χαρακτηριστικά γιατί δεν έρχεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι εσείς πιστεύετε ότι είσαστε ξεχωριστή χώρα σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη, στην Καταλωνία. Πάντως να θέσω κάποια από αυτά που είπατε σήμερα για τις πολιτικές που ακολουθήσατε στην Καλιφόρνια. Είπατε ότι απαιτείται να κερδίσουμε την ψυχή και την καρδιά των πολιτών. Πώς θα το κάνουμε αυτό όταν λέτε στις, ε, στους εκλογείς σας να δεχθούν ε, αυξήσει σημαντικότατες στους φόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του περιβάλλοντος. Λειτουργείται εις βάρος τους Συνεπώς υπάρχουν και άλλα θέματα τα, στα οποία οι φορολογικές σας πολιτικές και οι εμπορικές σας πολιτικές λειτουργούν εις βάρος των πολιτών. Όταν βλέπουμε εταιρείε όπως ο Elon Musk να παίρνει επιδοτήσεις κατά 4,9 δις από χρήματα των φορολογουμένων, προφανώς οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν θα έχουν μεγάλη τύχη. Εσείς προτείνετε στη πολιτική σας, στην πολιτεία σας, παρόλα αυτά 7,5 εκατομμύρια, 4 στους 10 είναι φτωχοί. 43% σύμφωνα με τις δικές σας στατιστικές των πολιτών δεν έχουν τους βασικούς πόρους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εσείς όμως συνεχίζετε να αυξάνετε τους φόρους και για το ε, περιβάλλον, αυξάνοντας έτσι τη φτώχεια. Οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν κυρίως τους φτωχούς, λέει ο ΣΑΣ και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Όταν λοιπόν το ίχνος του άνθρακα είναι ας πούμε 2,3 τόνοι για τους φτωχούς και 57% για τους πλουσίους, εσείς στην ουσία παίρνετε μέτρα στις Ηνωμένε Πολιτείες τα οποία χτυπούν φυσικά τους φτωχούς. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Έχετε καλές προθέσεις, θέλετε να προστατεύσετε το περιβάλλον, αλλά οι πολιτικές τις οποίε εφαρμόζετε βοηθούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχού, και οι φτωχοί θα υποφέρουν πολύ εξαιτία των πολιτικών σας. Λίζε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ Κυβερνήτα για μένα είναι πραγματικό προνόμιο ευκαιρία που έχω να μιλήσω εξ ονόματος ε, της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ομάδας μετά από τους δύο προλαλήσαντες. Δύο συνάδελφοι τώρα και στην προηγούμενη συνεδρίαση άλλος ένας είπαν ότι πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν με τον πρόεδρο Τραμπ. 500 εκατομμύρια είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορεί 10% των πολιτικών που εκπροσωπούν τους πολίτες αυτούς να συμφωνούν με τον Τραμπ. Και αν βρείτε 10% θα είναι και πολύ. Μπορεί να σας φανούν πολύ τα 50 εκατομμύρια, αλλά ουσιαστικά και, και οπωσδήποτε είναι μειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μειονότητα ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Πρόεδρος μας είναι ο Μάνφρετ Βέμπερ της κεντροδεξιάς ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και είπε όταν κυρώσαμε την ε, Συμφωνία των Παρισίων ότι είναι ε, η βασική υποχρέωση μας ε, και καθήκον για την επόμενη γενεά. Και όταν αποφάσισε ο Τραμπ να αποσυρθεί, ο Μάνφρετ Βέμπερ εξέδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε τώρα έχει έρθει η ώρα της Ευρώπης, η οποία θα πρέπει να αναλάβει την ηγεσία για να υποστηρίξει και να υπερασπιστεί αυτή τη συμφωνία γιατί είναι σωστή και γιατί εξασφαλίζει το μέλλον και του περιβάλλοντος και της βιομηχανίας μας. Και έκανε ρητή αναφορά σε εταιρείε και σε κράτη ε, και σε πολιτείες μάλλον των ΗΠΑ που συμμερίζονται την άποψη αυτή και τη δέσμευση, όπως είναι η Καλιφόρνια. Μπορείτε λοιπόν να διαβιβάσετε στι Ηνωμένε Πολιτείε ότι στην Ευρώπη το 90% των πολιτών και του πληθυσμού και των εκπροσώπων του συμφωνούν με τις δικέ σας απόψει. Όταν κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να υλοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή. Τι σημαίνει, στις 6 ακριβώς αρχίζει ο τριμερής διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων. Λοιπόν. Και θα αποφασίσουμε μέτρα που θα ενισχύσουν αυτό το σύστημα και όποιος επενδύει σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα θα κερδίσει. Όλα αυτά θα τα διαπραγματευτούμε σήμερα. Και στην προηγούμενη συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ακούστηκαν κάποιες ε, φωνές που διαφωνούν με τις φιλόδοξες προτάσεις για τα αυτοκίνητα. Η πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί καλή βάση για τη διαπραγμάτευση και για τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων στη συνέχεια. Θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή αγαπητέ κυβερνήτα σε ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε ήδη και από κάποιον άλλον ομιλητή προηγουμένω, που είναι η αεροπορία. Οι αερομεταφορέ έχουν μικρό μερίδιο σήμερα στι εκπομπέ, αλλά αν δεν δράσουμε αυτό θα καταβροχθήσει τις προσπάθειες που καταβάλουμε σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία για βελτίωση. Απογοητεύτηκα λίγο και από τη Χίλαρη Κλίντον όταν ήταν υπουργό Εξωτερικών γιατί οι προσπάθειες που έκανε η Ευρώπη δεν βρήκαν μεγάλη υποστήριξη στις ΗΠΑ. Χρειάζεται όμως συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, πιστεύω. Παρακαλώ προσέξτε το αυτό, διότι μπορεί να φαίνεται ίσονος σημασίας, αλλά αυξάνονται οι εκπομπές, διπλασιάζονται παγκοσμίω κάθε δεκαετία. Άρα χρειάζεται δράση από πλευρά μα και στο συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντάλη. Σας ευχαριστώ κύριε Μπράουν. Ήδη είχα την δυνατότητα να σας θέσω ερωτήσεις νωρίτερα και γι' αυτό θα είμαι συνοπτική. Γνωρίζω ότι όταν έχετε πολλές ερωτήσεις είναι δύσκολο να δώσετε απαντήσεις πλήρες. Απλά θα ήθελα να πω τις απόψεις μου για το COP23 και για τον ρόλο τον οποίο θα παίξουν οι πόλεις, οι περιφέρειες και οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία. Νομίζω ότι η COP23 είναι μια εξαιρετική ευκαιρία εάν πράγματι μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τις, ε, να υπάρξουν δράσεις για το περιβάλλον. Οι εθνικές παρεμβάσεις τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουν όλες οι χώρες μετά το Παρίσι πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Θέλουμε έτσι να αλλάξουν τα πράγματα και να αλλάξει η καθημερινότητα όλων. Για να συμβεί αυτό οι χώρες θα πρέπει να παρουσιάσουν τα εθνικά τους μέσα και να δείξουν το πώς θα μπορέσουν να επηρεάσουν τη μείωση των εκπομπών. Γνωρίζετε βέβαια ότι μετά την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτικών, Πολιτιών, συγγνώμη, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες στοχεύουν να κάνουν το ίδιο γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν το υψηλό τίμημα. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε τον βιομηχανικό κλάδο και τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα να ενδιαφερθεί και να δει ποιο είναι το συμφέρον του. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια του COP23 να συνεργαστούν, να είναι ένας χώρος συνεργασίας των βιομηχανικών ομάδων με τις πόλεις και τις περιφέρειες και θα πρέπει επίσημα το COP23 να αναγνωρίσει τις πρωτοβουλίες των περιοχών πολιτιών κτλ σαν τμήμα της δράσης εναντίον των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν σωστή συνεργασία από όλους τους εμπλεκομένους έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο βιώσιμη και αηφόρος οικονομία θέματα υπάρχουν στα οποία πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Οι κλιματολογικές αλλαγές δεν είναι απλό περιβαλλοντικό θέμα. Συνδέεται με την αποτελεσματικότητα και με την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Για να συμβεί αυτό απαιτείται καλή θέληση, απαιτείται πολιτική βούληση, απαιτείται σωστή θέσπιση και σεβασμός των στόχων όπως και μετά το Παρίσι απαιτείται με ενεργό τρόπο να αναζητήσουμε νέες ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Και νομίζω ότι όχι μόνο οι κυβερνήσεις μας, αλλά οι περιφέρειες μας, οι πόλεις μας, οι τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα θεωρήσουν ότι το COP23 είναι ένα καλό πλαίσιο για την προσπάθεια αυτή. Bilbao Barandica Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας σήμερα. Νομίζω ότι πραγματικά το να σας ακούει κανείς είναι σαν ένα ρεύμα φρέσκου δροσερού αέρα, ιδιαίτερα στα πλαίσια της πολιτικής για τις κλιματολογικές αλλαγές του Προέδρου σας πράγματι ο ρόλος των περιφερειών είναι σημαντικό. Εγώ είμαι Βάσκα και η κυβέρνηση της περιοχής μου από το 2016 έχει συνυπογράψει τη Συμφωνία COP21 ε, και παρόλα αυτά συμμετέχουμε πλήρως σε προγράμματα για τις κλιματολογικές αλλαγές, για τις συνέπειές τους. Εφαρμόζουμε λοιπόν και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα νέο πρότυπο το οποίο να είναι ένα αηφόρο συνεργαζόμαστε με τις ευρωπαϊκές αρχές έτσι ώστε να υπάρξουν αλλαγές στον τομέα του κλίματος έτσι ώστε να μην υπάρχουν απειλές εις βάρος του κλίματος αναφερόμενοι στη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης στο μέλλον δίνει την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αγαθών, ανακύκλωσης και έχει πάρα πολύ σημαντικές ε, συνέπειες για όλους μας. Δεν μπορώ τώρα να μπω σε περαιτέρω εξηγήσει. Υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Αλλά θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, έχουμε συζητήσει για το λεγόμενο fracking Νομίζω ότι και στο Κοινοβούλιο και σε διάφορες χώρες και σε διάφορες περιφέρειες. Τι γίνεται ακριβώς με αυτό το, το σχιστολιθικό αέριο. Έχουμε εργαστεί επίσης πολύ και για την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η άποψή σας είναι ότι μια εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν σε θέση να διευκολύνει τα μέτρα κατά πολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Εμείς υποστηρίξαμε την εμπορική αυτή συμφωνία, λόγω δυστυχώς όμως των πολιτικών αλλαγών που ενδιάμεσα συνέβησαν δεν υπήρξε μια τέτοια συμφωνία ουσιαστικά. Τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε στην καταπολέμηση των προβλημάτων που έχουμε από κοινού. Τώρα στις εμπορικές συμφωνίες τις οποίες έχετε εσείς με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, φαίνεται ότι θα υπογράψετε νέες συμφωνίες με την Ιαπωνία. Στοχεύετε στο να βελτιώσετε και να εντατικοποιήσετε τις σχέσεις σας με την Ινδία. Πιστεύετε ότι τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες ε, θα ε, βοηθήσουν ή θα οδηγήσουν σε αρνητικά βήματα για τα προγράμματα καταπολέμησης των κλιματολογικών αλλαγών. Και τέλος εσείς ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, πιο συγκεκριμένα, τι πιστεύετε για το ότι ο Ντόναλτ Τραμπ έχει βγει έστω και προσωρινά από τη Συμφωνία του Παρισιού. Θα ζητώ συγγνώμη, πρέπει να είμαι αλλού στις 6.30 δυστυχώς. Ο κύριος Εκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυβερνήτα Μπράουν. Είναι εντυπωσιακό ο απολογισμός σας ε, για την καταπολέμηση των εκπομπών αερίων ε, καυσαερίου και σας συγχαίρω. Θέλω να σας αναφέρω ορισμένα επιχειρήματα παράλληλα με αυτά που είπε η κυρία Χάζεκα. Θεωρώ ότι μία από τις κυριότερες ελλείψεις της συμφωνίας του Παρισίων είναι το ότι δεν λαμβάνει υπόψη η συμβολή της εκτινοτροφίας που υπολογίζεται στο 15 18% και επίσης ε, άρα είναι περίπου όσο και των μεταφορών. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να μειώσουμε μόνο τις εκπομπές καυσαερίου αλλά και άλλων αερίων όπως του μεθανίου που είναι 25% πιο επιβλαβές. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο διατροφής μας. Εάν αυξηθεί μέχρι το 2050 το 76, κατά 76% η κατανάλωση ε, κρέατος, ε, κάτι που θα γίνει αν δεν αλλάξουμε τις συνήθειές μας, τότε ε, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τεράστιες, ε, τεράστια κοπάδια που είναι υπεύθυνα για το μισό περίπου των εκπομπών μεθανίου. Τι κάνετε λοιπόν στο, στην πολιτεία της Καλιφόρνιας για να μειωθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις από την ε, παραγωγή κρέατος και ανάλωση κρέατος. Η Κίνα, για παράδειγμα, θέλει τα επόμενα 12-13 χρόνια να μειώσει και το τονίζω κατά 30%. Ίσως βέβαια ως αντιστάθμιση για το ότι η Κίνα χτίζει το ένα εργοστάσιο ηλεκτρισμού ε, με κατανάλωση άνθρακα ε, μετά το άλλο. Δεν θα ήταν λοιπόν δυνατόν εσείς που θα φιλοξενήσετε την επόμενη συνάντηση κλίματος στο Σαν Φρανσίσκο να προτείνετε κάτι εξίσου φιλόδοξο για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς την θέρμανση του κλίματος. Όπως λέμε, όποιος δεν μάχεται έχει ήδη χάσει τη μάχη. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τους συμπολίτε μας τι είναι πιο σημαντικό, η διατήρηση του πολιτισμού, όπως το γνωρίζουμε, είτε να φάνε άλλο ένα cheeseburger αυτό το ερώτημα πρέπει να έχουμε το θάρρος να το θέσουμε επιτέλους. Πώς αντιμετωπίζετε ε, αυτή την ε, πρόταση ε, κυβερνήτα Μπράουν, ο πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι 8 ομιλητές. Σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Θα είμαι συντομότατος. Μιλήσαμε πολύ για εκπομπές που είναι τμήμα της διαδικασίας. Πρέπει να μιλήσουμε όμως και για τις ε, επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα. 5 ε, δις κατέτος, ε, αν σκεφτείτε το τι ξοδεύουμε για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Είναι λίγοι αυτοί που είναι κατά δυστυχώς που δίνουν μάχη εναντίον των επιδοτήσεων αυτών. 1,5 δις η Γαλλία, 3,5 η Ιταλία, 5 η Γερμανία. Εσείς επενδύετε στις ανανεώσιμες και παρόλα αυτά όμως από τις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου εξακολουθούμε να εξάγουμε με απαράδεκτο τρόπο το πετρέλαιο. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε ότι εκεί που υπάρχει το πετρέλαιο δεν υπάρχει χρυσός μαύρος, υπάρχει φτώχεια και δυστυχία. Κοιτάξτε, παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι, γιατί στο τέλος θα είναι πολύ λίγοι οι βουλευτές που θα είναι παρόντες όταν δώσει απαντήσεις ο κυβερνήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Φλέξταϊν. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, κυβερνήτα Μπράουν. Εγώ ε, είμαι εξωτικό είδος εδώ, γιατί δεν ασχολούμαι με θέματα περιβάλλοντος, αλλά εξωτερικής πολιτικής και είμαι πρόσωπος ε, της ομάδας μου. Με ρώτησαν στο State Department ε, πριν από λίγο καιρό ε, τι θα γίνει αν αποχωρήσει ο πρόεδρος από τη Συμφωνία για το Κλίμα. Απάντησα τι θα συμβεί δεν ξέρω, αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η συναισθηματική απόσταση των πολιτών μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με άλλα πράγματα ε, που έχουν συμβεί στο τελευταίο διάστημα, με πιο πρόσφατη την ε, συμφωνία του Ιράν. Αυτό με απασχολεί και με ανησυχεί πάρα πολύ η συναισθηματική απόσταση, γιατί μεγάλωσα ε, τέλη της δεκαετίας του 50 ε, στο Βερολίνο και όποιος ε, έχει μεγαλώσει όπως εγώ εκεί έχει ένα δεσμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν μπορεί ποτέ να αλλοιωθεί. Αλλά παρόλα αυτά ε, εσείς που είστε υπέρ της κλιματικής αλλαγής, υπέρ του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών, υπέρ της θετικής νομοθεσίας Μα δείχνετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι μόνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πάρα πολλοί άλλοι πολιτικοί που συνεργάζονται μαζί μα και χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ. Κυρία Μπεθέρα. Ο κύριος Κόμπορν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπράουν, εδώ εμφανίζεστε ως αρχιερέας ε, που κάνει προσευχές ε, υπέρ της θρησκείας της ανθρωπομορφικής ε, κλιματικής αλλαγής. Αλλά η οικονομία μας χρειάζεται έναν Σαμψόν για να γκρεμίσει το ναό. Και ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο Σαμψόν. Οι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται περισσότερο για θέσεις εργασίας ε, και όχι για την κλιματική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή κανένα επιστήμονο δεν μπορεί να κάνει καμία μελέτη, να λάβει χρηματοδότηση για καμία μελέτη, αν δεν είναι υπέρ τη κλιματικής αλλαγής. Από ό,τι ακούσαμε όμως, ο σχετισμό αυτών των δύο δεν είναι τόσο σαφής. Και αυτό το έχει πει ο Πάτρικ Μου, ο πρώην πρόεδρος τη Greenpeace. Ορισμένοι βεβαίω ε, θα με καταγγείλουν που λέω ότι δεν έχουν αποφασίσει οι επιστήμονες αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά το 2007 το IPCC είπε ότι το σύστημα αυτό είναι μη γραμμικό και χαοτικό. Οπότε ε, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μακροχρόνιες προβλέψεις. Δεν είναι υπεροπτικό οι επιστήμονες να θεωρούν ότι μπορούν να μας τα λένε όλα. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε τέτοια πράγματα. Γιατί βλέπουμε ότι και στον ε, Άρη, για παράδειγμα, μειώνεται, μειώνονται οι παγετώνες, αλλά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στον Άρη. Μπορεί ε, βεβαίως να έχει να κάνει με πολλά πράγματα η μείωση των παγετών στην ε, γη, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο ε, με αυτό. Κοιτάξτε, η πλειονότητα δεν τα ξέρει όλα επειδή είναι η πλειονότητα. Εγώ ανησυχώ περισσότερο για το, τους ε, ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά στην ουσία βοηθάνε να ε, βγάζουν παραδάκι κάποιες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Μπράουν για την παρουσία σας. Δεν θα κάνω περισσότερες ε, ερωτήσεις. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Διότι Ξέρουμε πολύ καλά ότι η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε θύματα και οδηγεί σε επιπτώσεις για την ε, οικονομία. Η Ομοσπονδική Κυβέρνηση των ΗΠΑ χρειάστηκε να δώσει δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις. Το 2017 υπήρξε ε, τεράστιος ε, αριθμός καυσώνων παντού στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Πορτογαλία είχαμε την πιο ξηρή περίοδο των τελευταίων 10 ετών είχαμε τραγικές πυρκαγιές το καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο όπως και στην Καλιφόρνια εκατοντάδες χιλιάδες ε, στρέμματα έγιναν στάχτη καταστράφηκαν τα πάντα ζώνες προστατευμένες ε, εθνική δρυμή έγιναν στάχτη όπως είπα 5% της υπηρετικής Πορτογαλίας καταστράφηκε. Τέσσερις πόλεις κάηκαν. Είχαμε πάνω από 100 νεκρούς σε τέσσερις μήνες. Εκατοντάδες τραυματίες. 50% του, της οικονομίας μας από την υλοτομία καταστράφηκε. Το κόστος ε, υπολογίζεται σε πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι πέτρες δεν κάηκαν, λέμε, για τη χώρα μας. Όλα αυτά σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. και είναι κρίμα που ο πρόεδρος Τραμπ ε, αγνοεί το αυτονόητο. Ο αρμόδιος των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή είπε ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται όλο και περισσότερο. Και το περιθώριο που μας μένει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μειώνεται. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, πολύ ταχύτερα. Πρέπει να έχουμε περισσότερες φιλοδοξίες. Οπότε κύριε Κυβερνήτα Επαναλαμβάνεται συνεχώς ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι κοινή μας αποστολή. Και βεβαίως αυτό ισχύει. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες της Ευρώπης για να μειώσουμε τις δικές μας εκπομπές. Ενώ ε, μια χώρα που ε, μολύνει τόσο πολύ δεν κάνει τίποτα και συνολικά ε, επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και πολλοί αρνούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν την ε, συλλογική προσπάθεια, ενώ είναι αναγκαίο αν θέλουμε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Η 23η ΚΟΠ είναι βέβαια μια ακτίδα ελπίδας, οπότε σας ευχαριστώ για τη δέσμευση και την αποφασιστικότητά σας, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι ο πλανήτης μας δεν είναι μόνο η Washington. Πρέπει και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι μόνο η Washington. Πρέπει λοιπόν η αποφασιστικότητά σας ε, να βοηθήσει θα πρέπει να πείσουμε τον Τραμπ να αλλάξει γνώμη αλλά ας ελπίσουμε τουλάχιστον δεν θα πανεκλεγεί Μπριάνο Ευχαριστώ Πρόεδρε Κυβερνήτα, δύο είναι τα προβλήματα της εποχής μας, η μετανάστευση και το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι ο σωστός δρόμος είναι να χτίσουμε νέα τύχη και να αρνηθούμε την πραγματικότητα όπως το κάνουν ορισμένοι. Οι προκλήσεις αυτές και οι δυσκολίες και λόγω των, της μετανάστευσης που ξεκίνησε λόγω των κλιματολογικών αλλαγών υπάρχουν προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά τα οποία θα πρέπει να αντιμεταπιστούν με πολύ, πολλαπλό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη μας ε, την εφαρμογή της αρχής της ε, χωρίς όρια ανάπτυξης, των λίγων βέβαια, κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο οικονομικά και περιβαλλοντικά. Οι ευθύνες ε, του ανθρώπου είναι προφανείς όπως ακριβώς δείχνει και η τελευταία έκθεση του ίδιου του Λευκού Οίκου. Παρ' όλα αυτά ο Τραμπ αρνείται την πραγματικότητα και γι' αυτό η COP23 είναι μια καλή ευκαιρία. Και είναι μεγάλη χαρά μας που εσείς μαζί με άλλους ηγέτες τοπικούς προσπαθείτε να δείξετε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε η ένταση είναι υψηλή και η επιθυμία δράσης εξίσου υψηλή. Εμείς στην Ευρώπη ακολουθούμε τον δρόμο πλέον της κυκλικής οικονομίας, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την επανεξέταση της λειτουργίας της παραδοσιακής οικονομίας με νέα οπτική. Η κυρία Κιέγγε, πρόεδρε, κυβερνήτα, από τα παλιά χρόνια η ανθρωπότητα κινείται Πολλοί είναι αυτοί που μετακινούνται για να ψάξουν νέες ευκαιρίες, για να ξεφύγουν από διώξεις, για να ξεφύγουν από τη φτώχεια, για να ξεφύγουν από το κλίμα. Είναι οι λεγόμενοι κλιματικοί πρόσφυγες. Βλέπουμε τον κίνδυνο που υπάρχει στον Ειρηνικό με τα νήσους Βανουατού, με τα νήσους Φίτζι, όπου οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν άμεσα. Συνεπώς λοιπόν μετά από τη δήλωση της Νέας Υόρκης που υπεγράφησαν από τους διεθνείς ηγέτες πέρυσι στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών βλέπουμε ότι η σχέση της οικονομικής ανάπτυξης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι προφανής και αυτό επηρεάζει και την κινητικότητα των μεταναστών. Βέβαια δεν είστε εσείς αυτός τον οποίο θα πρέπει να πείσω αλλά ο πρόεδρός σας και νομίζω ότι στην ουσία αντιμετωπίζει με αρνητικό τρόπο αυτούς που έρχονται στις χώρες μας. Είναι άνθρωποι που διαφεύγουν από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και οφείλουμε να δίνουμε μάχη καθημερινή εναντίον της παραπληροφόρησης και θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μην αποδεχθούμε όπως και εσεί στην Καλιφόρνια τον αρνητισμό των συνεπειών στο περιβάλλον του Τραμπ βλέπουμε ότι η μετανάστευση συνολικά θα επηρεάσει ε, την εικόνα του κόσμου και θα υπάρξει και μία συμφωνία το Σεπτέμβριο του 2018 που θα μπορέσει να βοηθήσει να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Εύχομαι λοιπόν να πάει καλά η συνάντηση για το κλίμα την οποία οργανώνεται στην δική σας πολιτεία το επόμενο έτος. Τάνοκ. Ευχαριστώ. Εγώ συμμετέχω στην πλειοψηφία, λυπάμαι βαθιά που αποχώρησε από τη συμφωνία πρόεδρος Τραμπ, αλλά όπως είπες κάποιος μπορεί να μην επανεκλεγεί. Αλλά όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουμε πολύ καλά τις καταστροφικές επιπτώσεις που προβλέπονται για την υποσαχάρη Αφρική, για τις μεταναστευτικές πιέσεις και πρόσφατα στην Επιτροπή μου θα ψηφίσουμε για μια νέα έννοια του ε, κλιματικού πρόσφυγα που δημιουργεί πολλές διαφωνίες. Ξέρουμε ότι κάποια νησιά του Ειρηνικού μπορεί να βυθιστούν, αλλά δεν έχουμε ακούσει για τις αρνητικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ. Δεν αναμένεται επίσης να έχετε ισχυρότερες μεταναστευτικές πιέσεις από την Λατινική Αμερική. Δεν θα θυγεί η γεωργία σας, η δυνατότητά σας να συνεχίσετε να είστε στο βολόνας του κόσμου. Πώς θα μπορείτε να... Ε, αντικαταστήσετε την, ε, τις μορφές ενέργειας που έχετε τώρα με άλλες, θα χρησιμοποιήσετε την υδρορογμάτωση, θα χρησιμοποιήσετε τι για να παράγετε ε, ηλεκτρικό, γιατί έμαθα ότι είχατε και διακοπές πρόσφατα. Ε, να, μερικές ερωτήσεις ε, κύριε Κυβερνήτη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχετε το λόγο, όχι μόνο για δύο λεπτά φυσικά. Καλά, δεν με περιμένετε, περιμένετε από μένα τώρα να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Δεν έχετε εσείς αρκετό χρόνο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ε, τα κλιματιστικά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά και τα σπίτια μας πλέον είναι πολύ φιλικά προς το κλίμα. Έχουμε πλέον ε, ε, ε παθητική ε, αντανάκλαση ε, του ηλίου και ενέργεια που παράγεται κατά αυτόν τον τρόπο και πραγματικά έχουμε προοδεύσει πολύ στα κλιματιστικά. Ε, για τη μετανάστευση, η Καλιφόρνια έχει 25% ε, του πληθυσμού που έχει γεννηθεί σε άλλες χώρες. Πολλοί μεταναστεύουν στην Καλιφόρνια, ορισμένοι νόμιμα και άλλοι χωρίς άδεια. Παρόλα αυτά όμως, Ε, αυξάνεται ε, με ρυθμούς ε, πολύ μεγαλύτερους από ό,τι σε υπόλοιπες Ηνωμένε Πολιτείες η πολιτική νομοθεσία και για τη Γεωργία. Εσείς οι Βρετανοί είστε, έχετε καταπληκτική παιδεία και μιλάτε και τη γλώσσα του, τα, τα αγγλικά όπως μιλάει ο βασιλιάς η βασίλισσα αλλά τα κροκοδίλια δάκρυα που γίνεται για τους στοχούς δεν μπήθουν καθόλου μάλιστα Να το αποσύρετε αυτό λέει ο κύριος Βολφ το ε, πρόεδρος σας παρακαλώ πρέπει να σεβαστούμε τον προσκεκλημένο μας δεν μιλούσα σε εσάς κυρίως προς αυτή την πλευρά της αίθουσας, αλλά αν θέλετε σας συμπεριλαμβάνω και σας Ακούω διάφορα πυροτεχνήματα ρητορικά εδώ. Ε, και είναι πολύ δύσκολο να τα καταρρύψει κανείς ε, με έξυπνο τρόπο και, και λογικό. Πιο εύκολο είναι να πετάς πυροτεχνήματα παρά να απαντάς. Εδώ έχουμε την ποικιλομορφία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. μιλάτε, απαντούμε εμεί στι, Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, έχουμε και μεγάλες διαφωνίε και όποτε έχουμε τέτοιε διαφωνίε πώς τι λύνουμε με ψηφοφορία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν αποφασίζουμε και αυτή είναι η πρόκληση μπροστά μα γιατί υπάρχει μεγάλη διαφωνία. Ε, είπα και εγώ και άλλοι είπαν ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο για να κάνουμε όσα πρέπει. Και είναι πολύ σημαντικό και όσο και δύσκολο να σφυριλατήσουμε την απαραίτητη συνένεση για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά την αντίρρηση τώρα για τη σοβαρή ε, κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες ε, ε, μας λένε ότι πραγματικά είναι ανθρωπογενή σε μεγάλο βαθμό η κλιματική ε, αλλαγή. Μπορείτε να επικρίνετε την έκθεση της IPPC και να λέτε ότι είναι πληρωμένοι και δοτοί ε, και πουλημένοι επιστήμονες, αλλά αν δείτε οποιοδήποτε κατάλογο της επιστημονικής κοινότητας θα καταλάβετε ότι είναι και πραγματική κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις έχει. Και μεγαλύτερο αντίκτυπο θα έχει στο μέλλον, τα χειρότερα έρχονται. Μπορεί να μην σας πείσω γιατί εσείς ε, το βλέπετε από τη δική σας κοπιά και με μια πίστη, με πίστη σας. Και χαίρομαι που τα λέτε γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα και ποια είναι και τα προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο τον υπόλοιπο. Και γνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ είμαι επεπισμένος ότι οι επιστήμονες στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν δίκιο. Με μοντέλα, με μετρήσεις. Δεν χρειάζεται να επανέλθω τώρα για να σας παραθέσω όλα τα στοιχεία. Είναι πραγματικά συντριπτικά. Ακόμα και η κυβέρνηση Τραμπ ε, τελικά στην έκθεση της ε, παραδέχτηκε ε, τα αντίθετα από αυτά που λέτε και εσείς αναγκάστηκαν να βγάλουν μια επιστημονική έκθεση ακόμα και οι άνθρωποι του Τραμπ. Γιατί ε, ε, ε, ε, σοβαροί επιστήμονες, έγκριτοι, κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα με την Επιτροπή, αλλά ο κόσμος αυτά τα υποτιμά, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Και η άρνηση της ε, κλιματικής αλλαγής Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ το ανετικό και εδώ και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και όσο αυξάνει σε προσοχή και κερδίζει προσοχή, ο κόσμος πείθεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ότι ε, είναι πραγματικά ε, ζητήματα και προβλήματα κλιματική αλλαγή και υπερθέρμανση του ο πλανήτη. Τώρα για ε, τα γαλακτοκομικά, το κρέας και την κτηνοτροφία. Η παραγωγή μεθανίου από την κτηνοτροφία αλλά και από αλλού είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει πραγματικά να την αντιμετωπίσουμε το μεθάνιο, το βρώμικο άρθρακα και άλλες μορφές ε, ρήπανσης που έχουν βραχή βιομεν αλλά ρηπαίνουν πάρα πολύ. Θα πρέπει να μειώσουμε αυτούς τους βραχή ε, ρήπους και τις εκπομπές για να γίνει αυτό και όταν γίνει αυτό θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα να μιλάμε για χάμπουργκερ το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή δεν βοηθάει να επικεντρώνουμε σε κάθε μεμονωμένη πρωτοβουλία. Ε, είναι γενικότερη στόχοι. Ε, όταν έχει ένα γενικότερο στόχο, μειώνει ε, ε, ανατομέα τις εκπομπέ. Μεταφορές, ε, αερομεταφορές. Δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά. Ναυτιλία το ίδιο. Θα πρέπει με ένα συστηματικό τρόπο να το προσεγγίσουμε και γενικότερο, όχι επιμέρους τώρα τον κάθε κλάδο. Ο καθένας μπορεί να, να τρώει ό,τι θέλει. Αλλά αν συμφωνήσουμε και έχουμε πραγματικά εφαρμόσιμους στόχους που να μπορούμε να τους επιβάλλουμε ε, και υποχρεωτικούς και μειώσουμε τις εκπομπές με μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 ας πούμε ή νωρίτερα θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία ε, να δώσουμε στον καθένα την επιλογή. Τώρα δεν θα χρειάζονται ακραίες λύσεις ή απαγορεύσεις. Υπάρχει καινοτομία. Μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα με λιγότερο. Δηλαδή, ε, επειδή αυξάνεται η τεχνολογία, η πληροφορία σε σχέση με την πρώτη ύλη, μειώνεται η ποσότητα της πρώτης ύλης που χρειάζεται για να παραχθεί ένα προϊόν. Και έτσι μπορούμε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα με την καινοτομία, με την τεχνολογία, με τις επιστημονικές ανακαλύψεις. Επανέρχομαι στην Καλιφόρνια. Μειώνουμε τα αέρια του θερμοκηπίου. Έχουμε το πιο ε, πρωτοποριακό και επιθετικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και η οικονομία μας καλπάζει σε σχέση με ε, τον μέσο όρο. Ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες. 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έχουμε δημιουργήσει από την περασμένη οικονομική κρίση. Ε, με νέες γνώσεις, ε, με νέα στοιχεία μπορούμε να περιορίσουμε το αποτύπωμα που αφήνει ο άνθρωπος ο ίχνος στο πλανήτη. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη και φεύγουν χρειάζονται μεγάλη συνένεση. Με δημοκρατικό τρόπο δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα σε κανέναν Εάν είμαστε τυχεροί και τα καταφέρω. Βεβαίως και το διοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει να ε, ε, ε, περιοριστεί. Για τα θέματα του εμπορίου υπάρχουν διαταραχές στο εμπόριο. Ας πούμε 20-30 δολάρια πληρώνονται οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητομηχανία, στην πετρελαιοβιομηχανία στι Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ στο Μεξικό είναι μισά τα ημερομίσθια. Δεν χρειάζεται να ορθώσουμε φραγμούς και εμπόδια, αλλά ένα κόσμο που να είναι στην υπηρεσία όλων μας. Αυτοί που λένε μην κάνεις τίποτα για την κλιματική αλλαγή, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, οι πλούσιοι, αυτοί που συνεδριάζουν σε τέτοιες αίθουσες. Όχι, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα υποφέρουν και θα πληγούν. Ο κοινωνικός αντίκτυπος θα αυξήσει τις διαφορές και θα ανοίξει η ψαλίδα ακόμα περισσότερο ανάμεσα σε πλουσίους και φτωχούς. Μην κάνουμε λάθος. Οι συνέπειες θα έχουν τεράστια σημασία και ως προς τον πολιτισμό στις κοινωνίες μας ε, θα είναι λιγότερο εύκολο να διοικούνται και θα έχουμε και τις επιπτώσεις της υπερθέμασης του πλανήτη. Μειωμένη παραγωγικότητα στη γεωργία, ε, αύξηση του επιπολασμού των τροπικών νόσων, αύξηση της στάθμης των ωκεανών. Αυτά συμβαίνουν ήδη. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν το θερμότερο από ότι έχει καταγραφεί ποτέ. Αυξάνεται η θερμοκρασία. Και μπορεί και το 2 να είναι πολύ, ίσως 1,5 να είναι το όριο βαθμούς Κελσίου. Μιλάτε για βεβαιότητα. Εκεί να δείτε βεβαιότητα. Ορισμένοι λένε ότι δεν πιστεύουμε τους επιστήμονες, παίρνουμε φόρα και τραβάμε μπροστά και μετά τι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Η εξουσία ισχύει στον ανθρώπου της νανοτεχνολογίας, ε, γενετική μηχανική, ε, πυρηνική τεχνολογία, ε, πυρηνικά όπλα, όλα αυτά. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ ισχυροί, έχουμε δισεκατομμύρια αυτοκίνητα ενώ πριν από χρόνια είχαμε 300 εκατομμύρια. Έτσι ε, ε, ε, αυξάνεται η καμπύλη της εξουσίας που μπορεί να είναι καταστροφική και ολέθρια κάποια στιγμή. Απ' την άλλη υπάρχει και η καμπύλη πέρα από εκείνη της εξουσίας, της αυτοσυγκράτησης, της λογικής, της φρόνησης που είναι τελείως ευθεία και ο από τις Ηνωμένε Πολιτείες, μάλλον από τη Μεγάλη Βρετανία, ε, ε, λέει ότι η ανθρωπότητα έχει περίπου 50% στην καλύτερη περίπτωση πιθανότητες να επιβιώσει το 21ο αιώνα. Και θα πρέπει κάθε μονομένη δράση να αναλυφθεί και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χρειάζεται συνένεση, πρακτικά βήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Η COP23 ε, είναι το επόμενο σημαντικό βήμα Ήμουν στο Ρίο το 1992 όταν άρχισε να γεννιέται αυτή η προσπάθεια με μεγάλη αισιοδοξία και με όλα αυτά τα χρόνια μετά ακόμα διαπληκτιζόμαστε, ακόμα αγωνιζόμαστε, ορισμένα κράτη αδρανούν και τα επιστημονικά δεδομένα και η γνώση εξακολουθεί να τα υποστηρίζει αυτά. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι το μόνο μας πρόβλημα. Όπως γνωρίζετε, δύο λεπτά χρειάζεται για να φύγει μια πυρηνική βόμβα και να δρομολογήσει ποιος ξέρει τι και να πυροδοτήσει. Μπορούμε να παράγουμε τόσο πλούτο που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια αυταρέσκεια και συγκατάβαση ότι όλα είναι καλά και ωραία γιατί όλα είναι ωραία εδώ μέσα. Όχι, έχουμε, είμαστε σε μια πορεία, σε μια τροχιά καταστροφική χωρίς γυρισμό. Το βήμα το σημαντικό έγινε με το COP21, ήταν θετικό και νομίζω ότι το COP23 είναι το επόμενο βήμα και μετά το COP24 κτλ. Η έκκληση που απευθύνω λοιπόν εδώ είναι να πάρουμε σοβαρά τις επιστημονικές απόψεις να σχεδιάσουμε σωστά και με λογικό τρόπο το επόμενο βήμα και αν το πετύχουμε αυτό τότε θα κάνουμε τον κόσμο να δουλεύει καλύτερα από ό,τι σήμερα. Και ο κόσμος αυτός θα πάει καλά να ακολουθήσουμε τις συστάσεις αυτών που λένε ξεχάστε το δεν έχουμε πρόβλημα, δεν θα ισχύσει αυτό βέβαια. Έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας, τεράστιο πρόβλημα, έχουμε λύσεις, χρειαζόμαστε σημαντικές τεχνολογικές προόδους, συστοιχίες μέτρων και στον τομέα των αυτοκινήτων που θα πρέπει να είναι φθηνότερα και να καταναλώνουν λιγότερο από ό,τι σήμερα. Παντού λοιπόν μπορούμε να δράσουμε. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες στις οποίες να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για διασκέδαση, για τις ε, ομάδες, τον αθλητισμό, αλλά στην ουσία αγνοούμε για το περιβάλλον, ενώ εδώ υπάρχει ένα επίπεδο γνώσης και ευθύνης ικανό να βοηθήσει την κατάσταση. Η έκκληση που απευθύνω λοιπόν είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε την πράσινη δράση με την οικονομική πρόοδο. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς επιστημονική γνώση, χωρίς σοφία επιστημονική και χωρίς στενή συνεργασία. Κάνετε πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερα από ό,τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, ίσως όχι πιο πολλά από ό,τι κάνουμε εμείς στην Καλιφόρνια, αλλά όλοι μαζί από κοινού μπορούμε να κάνουμε πολλά, να δεχθούμε την αλήθεια, να παραδεχθούμε την αλήθεια, να συνειδητοποιήσουμε τα προβλήματά μας και να μην ξοδεύουμε χρόνο στις ανοησίες οι οποίες ακούγονται δεξιά και αριστερά. Λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε απαθείς, δεν μπορούμε να είμαστε αδρανεί πρέπει με φάνταστο τρόπο να αντιδράσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κομβικός παίκτη και θα επηρεάσει το αν πετύχουμε ή όχι. Όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ήρθα λοιπόν εδώ γιατί ήδη κάνετε πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν συμφωνούμε όλοι για το τι πρέπει να γίνει, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίσει η πρόοδος και να μην αποθαρρυνθούμε γιατί δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα των προσπάθειών μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρούμε λύσεις και λύσεις θα βρεθούν. Πρέπει με πολιτικό τρόπο θα πρέπει να κερδίσετε τις απόψεις των εκλογών, εκλογέων σας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Πρέπει να έχουμε πειθό και να πείσουμε και τον εαυτό μας να κάνουμε ακόμα απεραιτέρω ε, βήματα. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Χρειάζονται περισσότερα και είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα. Υπάρχουν ισχυρότατοι άνθρωποι εδώ που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για να έρθει στο σωστό δρόμο ο κόσμος και να μείνει στο σωστό δρόμο. Κοιτάξτε, έκανα λάθος, είναι και ο κύριος Πέτερλε εδώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κυβερνήτα, θέλω μόνο να σας συγχαρώ. Να σας συγχαρώ για τη συμμαχία, για το κλίμα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρο ότι θα ισχύσει, θα ενισχύσει την διατλαντική συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε. Ε,